συνεδρίασης. Τώρα θα έρθουμε στο πρόγραμμα της συνεδρίασης για αυτή την εβδομάδα από διάσκεψη των Προέδρων βάσει του άρθρου 59 ε, ε, του κανονισμού ε, εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη για σήμερα δεν υπάρχουν προτάσεις τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης. Για την Τετάρτη το απόγευμα μου είπαν, ε, μου πρότειναν το εξή, προτάθηκε το εξή. Και μάλιστα από του συντονιστέ τη ομάδα, η έκθεση τη κυρία Λούνερ για τι συμφωνίε σύνδεση και σταθεροποίηση για το κοσυφοπαίδιο και η δήλωση τη Αντιπροέδρου για τι ε, συστηματικέ ε, θανατώσει θρησκευτικών μειονοτήτων θα διαπραγματευτούν στην εξή σειρά. Πρώτα κοσυφοπαίδιο και μετά μαζικές θανατώσει Μετά την διακήρυξη της Αντιπροέδρου και είπα τη εκπροσώπου για τις ε, συμφωνίες σύνδεση με Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία και θα συμπληρωθούν στην ημερήσια διάταξη. Έχετε καθόλου αντιρρήσει εάν όχι, ε, αποφασίζονται, ε, αποφασίζεται ω και εγκρίνεται το πρόγραμμα εργασία. Παρακαλώ κύριε Λάμπερ. Πρόεδρε, πριν εγκρίνουμε τη μέρη διάταξη, θα ήθελα να πω το εξή. Στην διάσκεψη των Προέδρων συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα το θέμα τη Δανία. Η κατάσταση αυτή είναι εξαιρετικά ανησυχητική γιατί κάποια μέτρα θα σε αυτές τις χώρες τα οποία ε, ε, στα μάτια πολλών μελών ε, συνιστούν παραβιάσεις. Λεπάμε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Λέω Μιλτής, περιμένετε, λέει ο πρόεδρος. You Θέλετε να συνεχίσω στα αγγλικά. Όχι ε, στα γαλλικά, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε κατά πόσο γίνεται διερμηνία στα γαλλικά να, μπορούμε να ζητήσουμε τους διερμηνείς από τα αγγλικά να μεταφράσουν τα δικά μου αγγλικά σε ορθά αγγλικά. Όχι, υπάρχει διερμηνία στα γαλλικά. Ωραία, λοιπόν. Η κατάσταση στη Δανία πραγματικά είναι ανησυχητική υπό την έννοια ότι λαμβάνονται κάποια μέτρα των οποίων έχει προβλεφθεί η τελική έγκριση στις 26 Ιανουαρίου, μέτρα τα οποία σε ορισμένου από εμά ε, ε, φαίνεται ότι αντιβαίνουν στις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητήσαμε αυτό στη διάσκεψη των Προέδρων και συμφωνήσαμε για μια διαδικασία η οποία είναι εξή ότι σήμερα η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ε, περιμένει, αναμένει έναν, από ένα εκπρόσωπο της δανικής κυβέρνησης και μετά από αυτή τη συνάντηση θα συνέλθει η Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών και θα αποφασίσει κατά πόσο ε, χρειάζεται να γίνει μια συζήτηση στην Ολομέλεια γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμη ε, κατά πόσο η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα ε, γίνει αυτή η ακρόαση με τον ε, εκπρόσωπο της κυβέρνησης δεν θα γίνει σήμερα το βράδυ και αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι οι συντονιστές ε, δεν θα συναντηθούν σήμερα. Άρα λοιπόν στο πλαίσιο αυτό θεωρώ φυσιολογικό κύριε Πρόεδρε να προβλέψουμε ένα χρονικό διάστημα στην Ολομέλεια για να συζητήσουμε για την κατάσταση στη Δανία γιατί δεν γνωρίζουμε κατά πόσο η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα αποφασίσει να συνεδριάσει με ένα εκπρόσωπο της ανικής κυβέρνησης. Εάν δηλαδή ε, ε, γίνει αυτή η σύντηση θα γίνει εκ των υστέρων. Δηλαδή ε, στην, Ολομέλεια, στην πρώτη Ολομέλεια του Φεβρουαρίου, αλλά θα είναι μετά από την απόφαση της δανεικής κυβέρνησης. Άρα λοιπόν, κατανοώ πλήρως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αποφανθεί παρά επί αποφάσεων ε, νομοθετημάτων τα οποία έχουν ε, υιοθετηθεί στις χώρες μέλη και έχει την έννοια της προειδοποίησης. Άρα λοιπόν ε, θα είχε περισσότερο νόημα να γίνει αυτή η συνεδρίαση πριν και όχι μετά, όχι εκ των υστέρων. Και εγώ θεωρώ ότι εάν τελικά η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών συνέλθει και το ίδιο και οι συντονιστές, τότε η συζήτηση αυτή θα γίνει στην ε, Ολομέλεια. Ευχαριστώ κύριε Λάμπερτς. Νομίζω είναι σαφές. Σήμερα πληροφορήθηκα ότι η Επιτροπή Ελευθεριών θα συζητήσει, δεν θα συζητήσει το θέμα αυτό απόψε. Ζήτησα κατόπιν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να προβλέψει μια συνεδρίαση της Επιτροπής αυτής αύριο. Ε, είμαι διατεθειμένος ανά πάση στιγμή αύριο να μπορέσουμε κάτω εξαίρεση να ακούσουμε τα, αποτελε... τα συμπεράσματα της Επιτροπής. Στην περίπτωση που ζητηθεί η συζήτηση στην Ολομέλεια. Αντιλαμβάνομαι πως η Επιτροπή έχει πάρα πολύ γεμάτη ημερήσια διάταξη σήμερα, αλλά δεδομένη της απόφασης διάσκεψης των Προέδρων ζήτησε από τον κύριο Μόραες να προβλέψει τουλάχιστον μια συνάντηση των συντονιστών αύριο. Τρέψατε μου μια διευκρίνηση. Πρόκειται για μια συνάντηση των συντονιστών είτε όλη τη Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών, παρουσία ενό εκπροσώπου τη Ανική Κυβέρνηση. Ναι, κύριε Λάμπερτ. Κοιτάξτε, ε, ε, δεν έχει νόημα να γίνει συνεδρίαση χωρίς εκπροσώπους της ε, κυβέρνησης Δανίας. Τι θα συζητήσουν. Τηλεφώνησα στον Πρωθυπουργό της Δανίας και του ζήτησα να αποστείλει κάποιον εκπρόσωπο. Ο κύριος Βέμπερ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να στηρίξω το έτοιμά σας το διαδικαστικό, δηλαδή να ελέγξουμε την ε, νομική κατάσταση. Τώρα, να πω το εξής. Εάν σε κάθε περίπτωση εθνικής νομοθεσίας έχουμε τέτοιο εκνευρισμό και τέτοια κινητοποίηση όπως τώρα αυτή που κάνουν οι πράσινοι πραγματικά θα βλάψουμε την ε, ευρωπαϊκή υπόθεση. Πρέπει να σεβαστούμε τους δανούς συναδέλφους. Αυτοί πρέπει πρώτα απ' όλα να διαμορφώσουν την νομοθεσία τους ε, περί ασύλου και μετά μπορεί να τη συζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ομάδα μου δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάτι το κατεπήγον. Η κυρία Τσίμερ. Κύριε Πρόεδρε. Και εγώ στηρίζω την διαδικασία την οποία προτείνεται και βασίζομαι στο ότι αύριο θα έχουμε κάποια πληροφόρηση. Στον κύριο Βέμπερ θα ήθελα να πω το θέμα δεν είναι κάποιο προηγούμενο εδώ πέρα ή κάποια κανονική νομοθετική διαδικασία. Το θέμα είναι το εάν ε, θα συνεχίσουμε να σεβόμαστε τα, τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και σε αυτά ανήκει το δικαίωμα του ασύλου και όχι το να κατάσχονται τα τιμαλφή των προσφύγων. Μάλιστα νομίζω ότι συμφωνούμε. Θα μιλήσω ξανά με τον κύριο Μωραές για να υπάρξει μια συνεδρία σε αύριο. Ωραία. Λοιπόν, για την ημερήσια διάταξη. Τίποτα άλλο? Όχι. Κύριε Μαριά, για την ημερήσια διάταξη. Αργότερα λοιπόν. Καλώς. Περνάμε λοιπόν στο σημείο της έκθεσης Λάγκινε, της έκθεσης και την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον λόγο έχει ο εισηγητής. Wer übernimmt jetzt? Äh,